επόμενο θέμα η έκθεση του κυρίου Μπόρις για την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η αξιολόγηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων γίνεται για πρώτη φορά. Η έκθεση την οποία έχω καταρτήσει είναι μια έκθεση που αναλύει την κατάσταση. Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύω αυτή τη οδηγία. Είναι θετική εν γέννη αυτή η αξιολόγηση, ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την έκθεση με κάποιους μήνες καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα ήταν καθυστερήσεις ε, στην υλοποίηση από πλευράς κρατών μελών. Όπως τονίζεται όμως πλέον όλες οι χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει αυτή την οδηγία και αυτό συνιστά μεγάλη επιτυχία. Διότι εν λόγω οδηγία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ελευθεροτυπία αλλά είναι και ένα μέσο για την ε, εγγύηση της επιλογής, ε, στο, της ελευθερίας επιλογής στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ρυθμίζεται η κατάσταση αυτή. 8.000 είναι οι οπτικοακουστικοί φορεί σήμερα. Και υπάρχουν και άλλες 2.000 ε, συνδρομητικοί φορείς. Ε, η διαφήμιση επίσης ρυθμίστηκε, 12 λεπτά είναι ο κανόνας και θα πρέπει να διατηρηθεί. Ο κανόνας επίσης ε, περί χώρας προέλευσης είναι ένα σημαντικός κανόνας. Αν ο φορέας οπτικοακουστικός τηρεί κάποιες ε, απαιτήσει σε μια χώρα, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε μια άλλη χώρα. Αυτός είναι ένας πολύ καλός κανόνας. Είμαι μέλος Επιτροπής Πολιτισμού και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά επηρεάζονται από τις διαφημίσεις. Θα πρέπει ανήλικοι λοιπόν να προστατεύονται από διαφημίσεις ενοπνευματοδών, τσιγάρων και διαφόρων ε, τροφίμων ανθυγινών. Επίσης, ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι κάτι που ε, αναφερόταν και στην προηγούμενη έκθεση ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, ε, εφαρμόζεται. Παρότρινση ε, σε μίσος ήταν ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε έναν τηλεοπτικό σταθμό που αναφέρεται ως παράδειγμα που είναι αντισημιτικός, αντισημιτικό περιεχόμενο πρόβα προέβαλε. Επίσης τα ευρωπαϊκά δημιουργήματα τα προστατεύουμε Ευρωπαϊκά είναι το 63% των προγραμμάτων και 33% από ανεξάρτητους παραγωγούς. Είναι κάτι που το χρωστάμε και στην οδηγία. Αλλά θα ήθελα να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην πρόθεση των ευρωπαϊκών έργων τέχνης και δημιουργημάτων. Η οδηγία επίσης ζητά καταπολέμηση της ε, διακριτικής μεταχείρισης ε, λόγω ηλικίας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Ή επίσης ε, τι γίνεται με τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι βαρύκο ή μπορεί να είναι τυφλή. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Θέλουμε να συνεχιστεί η προσπάθεια και θέλουμε να ληφθεί υπόψη στο μέλλον και η περίπτωση της υβριδικής τηλεόρασης. Δεν κάνουν διάκριση αυτή τη στιγμή οι κατάλληλες μεταξύ επιγραμμικών και μη υπηρεσιών. Θα πρέπει όμως ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις εξέλιξεις τεχνολογίας στην τη τηλεόραση. Ίσως θα μπορούσαμε μετά από κάποια χρόνια να επανεξετάσουμε την οδηγία, αφού όμως παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, που βοήθησαν και προσβλέπω και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. σε ευχαριστώ πολύ. Πρώτος ομιλητής είναι ο κ. Παπα-Νικολάου. Κύριε Πρόεδρε, Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τον εισηγητή μας και να τον ευχαριστήσω γιατί κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του τελικού κειμένου απεδέχθη και τις τροπολογίες μας, των περισσότερων από εμάς και ήταν υπόδειγμα ε, συνεργασίας όλη αυτή την περίοδο. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο άρθρο 6 της οδηγίας ε, στο οποίο υπάρχει η πρόβλεψη της απαγόρευσης της υποκίνησης σε μίσος για λόγους φυλής φύλου θρησκείας ή εθνικότητος. κάνω ειδική αναφορά σε αυτό κύριε πρόεδρε γιατί βιώνουμε όλη μια περίοδο που η ακραία ρητορική βρίσκει έφορο έδαφος σε πολλά κράτη μέλη και πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι υποκινούν τέτοιες ακραίες τοποθετήσεις ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται με βάση το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο αυτής της οδηγίας που την έκθεση για πρώτη φορά επεξεργαζόμαστε σήμερα για την ενσωμάτωση και την εξέλιξή της και πρέπει όλοι εκείνοι που έχουν τέτοιες διαθέσεις να γνωρίζουν ότι ε, υφίσταται έλεγχος αυστηρός της Επιτροπής και κάθε φορά που θα προκύπτει παράβαση αυτό και θα ελέγχεται και θα, ε, θα, θα υπάρχουν κυρώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρα πολλού ε, ομιλητές από το ΕΛΚ. Κανονικά όταν έχει πάρει κανείς το λόγο δεν ξαναμιλάει σε αυτές τις συζητήσεις. Κυρία Μπαζέσκου, πρώτα. Κυρία Σερένσκα, να μιλήσουν για την ομάδα. Κυρία Μπαζέσκου, πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία για τις υπηρεσίες της οπτικοακουστικές είναι ένα βασικό στοιχείο του κανονισμού, της νομοθεσίας στον τομέα στην Ένωση. Θα ήθελα όμως η δημόσια διαβούλευση για ενδεχόμενα θεώρηση οδηγίας να είναι ευρύτερη. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στην ανεξαρτησία των εθνικών φορέων, ρυθμιστικών φορέων στα κράτη-μέλη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το άρθρο 9, παράγραφος 2, που ενθαρρύνει τα μέσα ενημέρωσης να θεσπίζουν δεντολογικούς κώδικες σε άλλους τομείς, εκτός του εμπορικού. Πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου περί ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και περί πλουραλισμού. Αναφέρεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εποπτικοί μηχανισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίοι θα ελέγχουν τις εξελίξεις στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και θα μπορεί τελικά φορέας να δίνει συστάσεις. Ευχαριστώ κυρία Σάντσε Σμιτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα κείμενο που ήταν φιλόδοξο για να πλαισίσει τα στηριότητα των οπτικοκουστικών μέσων ενημέρωσης και φαίνεται ότι ήταν κάτι επιτυχές απαιτείται μεγαλύτερη προστασία στα έργα τα ευρωπαϊκά, προστασία μεγαλύτερη των ανηλίκων, προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφία, όριο όσον αφορά και τις πολλές διαφημίσεις. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επί παραγράφου 13 της εκθέσεως Μπορείς. Εκεί ζητείτε ρητά οι υπηρεσίες, οι οπτικοκουστικές και τα μέσα ενημέρωση να εξαιρούνται από κάθε εμπορική συμφωνία. Ψηφίζουμε την Πέμπτη την εντολή για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τις ΗΠΑ. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι συνεκτικό στα και να ζητήσει και ρητή εξαίρεση των εκουστικών υπηρεσιών που να είναι εκτός των εντολών της διαπραγμάτευσης. Μια συμφωνία που θα συμπεριλάμβανε αυτές τις υπηρεσίες θα υπονόμευε τη μελλοντική βελτίωση της, της διοδηγίας που συζητούμε σήμερα. Αν δεχτούμε την απελευθέρωση του τομέα, απειλούμε την πολιτισμική ποικιλομορφία που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, θεμελιώδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα πρέπει να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό και, την και τα ευρωπαϊκά οπτικοκουστικά μέσα έναντι των ΙΠΑ. Ε, Ευχαριστώ. Η κυρία Σιλεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτή η έκθεση εστιάζεται επί πολλών σημαντικών ζητημάτων και χαίρομαι που εισηγητής ο κύριος Μπόρις αποφάσισε να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που έχουν προβλήματα ακοής ή όρασης. Η τηλεόραση είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά τώρα διαδίδεται και στις ε, φορητές συσκευές μας. Υπάρχουν άτομα όμως με αναπηρία που χρειάζονται και άλλες υπηρεσίες, όπως ε, νοηματική γλώσσα, να έχουν πρόσβαση στη νοηματική γλώσσα. Η προσφορά μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ευρύτερη, να καλύπτει και τις ανάγκες και αυτών των ανθρώπων, γιατί έτσι θα καταργηθούν πολλοί φραγμοί που υπάρχουν ακόμα στις κοινωνίες μας. Είμαι σίγουρη ότι θα συμβάλλει κάτι τέτοιο και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από τον οποίο υποφέρουν καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Ο κ. Ματούλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων, η ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης ε, έχει γίνει προτεραιότητα. Ελευθερία πρόσβαση, ε, πληροφορία, ελευθερία έκφρασης, εμπορικές πτυχές. Όλο και περισσότεροι λόγω του διαδικτύου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οπτικοακουστικού τομέα, παραδοσιακές και μη. Η συμπεριφορά λοιπόν των καταναλωτών, η αγορά μεταβάλλονται συνεχώς. Η αναγκη της Κομισιόν για την εφαρμογή των ε, υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων είναι σημαντική γιατί στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να προσαρμογή των κανονισμών. Ίσως ε, ε, καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να πάρουν και άλλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων ε, ε, από διαφημίσεις που προωθούν ανθυγινό ε, τρόπο διαβίωσης, μεταξύ άλλων ανθυγινά τρόφιμα, λιπαρά κτλ. Επίσης προώθηση των ανεξάρτητων έργων, 10% προβλέπεται, μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είναι σημαντικό να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτές και τα άτομα με προβλήματα όρεσης ακοής. Ευχαριστώ. Κυρία Κρούς, έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Αν έχετε λάβει το λόγο μια φορά σε αυτές τις συζητήσεις δεν μπορείτε να ξαναπάρετε το λόγο. Δεν ακούμε τον ομιλητή. Νομίζω ότι κάνετε διάκριση για το ΕΛΚ, λέει ο μιλητή. Ωραία, κατ' εξαίρεση θα σα δώσω το λόγο, λέει ο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στις αρχές, γιατί πήραν το λόγο μόνο ομιλητές από το ΕΛΚ. κατάλαβα ότι περασμένη φορά θεωρήσατε ότι καταχράστηκα του χρόνου μου Α, τώρα όμως θα σας ε, ε, απογοητεύσω ίσως τώρα να, θα είμαι σύντομος Συμφωνούμε με την έκθεση Μπόρις το σημείο 7 το σημείο 9 το, στο σημείο 17 είμαστε 100% σύμφωνοι η έκθεση αυτή πρέπει να υποστηριχθεί λοιπόν και τέλειωσα και πριν από το χρόνο που μου είχατε δώσει πρόεδρε τώρα επίτροπε Κρούς λέει ο πρόεδρος έχετε το λόγο θα ήθελα να πω πρώτα πρώτα ότι δεν είμαι από το ΕΛΚ Παίρνω τον λόγο λοιπόν και λέω ότι η έκθεση Μπόρις είναι πάρα πολύ καλή. Χαιρόμαστε, θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις μελλοντικές της δράσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Η Κομισιόν θα ξεκινήσει ένα, μια μελέτη για την προστασία των ανηλίκων από τις διαφημίσεις συνοπνευματοδών. Τα αποτελέσματα πρέπει να τα έχουμε μέσα στο 2013. Επίσης, ε, εκδώσαμε μία πράσινη βιβλό για τη σύγκληση και πραγματικά μιλάμε και για διάφορες κοινωνικές ομάδες που, των οποίων η άποψη πρέπει να ακουστεί και οι ανάγκες να καλυφθούν. Πάντως κύριε Πρόεδρο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει ε, πολλές από τις νέες λειτουργικότητες δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη ή δεν χρησιμοποιούνται ακόμη αλλά σίγουρα έχει προχωρήσει τεχνολογία και ε, την οποία χαιρετίζουμε η οποία υπάρχει και την πράσινη βίβλο αναφερόμαστε ακριβώς σε αυτό το θέμα τι, θα πρέπει, τι πρέπει να κάνουμε και μετά τα πορίσματα από τη διαβούλευση για την πράσινη βίβλο θα και κάνουμε προτάσεις για συγκεκριμένα, συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένε δράσεις. Μιλούμε εδώ για τηλεοράσει με ενσωματωμένε υπηρεσίε, διαδικτύου αν μπορώ να το πω έτσι. Αυτές, αυτή είναι η καινούρια τεχνολογία για την οποία μιλούμε και βεβαίω πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τι ανάγκε των ορισμένων κοινωνικών ομάδων, την προστασία για των ανηλίκων για τα χρηματοδοτικά ε, μοντέλα, υποδομές, ε, ε, καθεστώτα ιδιοκτησίας κτλ. Και εδώ μπαίνουμε στα χωράφια στα οποία μπαίνει και η πράσινη βίβλος ε, της ελευθεροτυπίας που συζητούσαμε προηγούμενα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του και την ε, Επιτροπή Πολιτισμού επίσης Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Αύριο η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση της κυρίας ε, Ρία Όμεν Ρόιτεν για τις συντάξεις. Θέμα που υποσχολεί όλους μας φαντάζομαι. Κυρία εισηγήτρια έχετε το λόγο. Voorzitter, geachte Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Κρούζ, χαίρομαι που είστε εδώ παρούσα. Θα ήθελα να ξεκινήσω